Κυρίε και κύριοι, άρχεται η συνεδρία τη Επιτροπή Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη. Προηγουμένω συνεδρίασαν οι συντονιστέ και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 2, την έγκριση τη σα διάταξη. Έγκριση των πρακτικών τη προηγούμενη συνεδρίασης. Έχουμε και απευθείας μετάδοση με βάση την πρόταση για τα νέα τρόφιμα της κυρίας Άρβου έχουμε αλλαγή το σημείο της ημερήσιας διάταξης και το σημείο 7 θα το συζητήσουμε μετά το σημείο 9. Έχουμε διερμηνία από και προς γερμανικά, γαλλικά, Η κυρία Σάιερ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε εγκρίνει ήδη την ημερήσια διάταξη γιατί είστε πολύ γρήγορος και δεν σας προλαβαίνουμε. Αν δεν υποβληθούν ε, παρατηρήσεις ε, για τα πρακτικά θα θεωρηθούν συγκεκριμένα. Το είπαμε αυτό. θέλετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, στο σημείο 18 έχω κάποιες παρατηρήσεις. Έγινε εκτενή συζήτηση, ενδιαφέρουσα. Πολύ καλό το ψήφισμα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι μέλη από εδώ και πέρα. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να δώσουμε ίση προσοχή σε όλους τους τομείς και του βόηου κρέατος, του χείριου. Θα πρέπει όλοι οι τομείς να τύχουν της δέουσας προσοχής. Και επίσης θα πρέπει να στηριχτούμε στο ψήφισμα, να δούμε τα μέσα και τα κονδύλια που έχουμε μέσα των διαθροτικών ταμείων αλλά και των άλλων ταμείων. Ευχαριστώ. Πολύ σωστά. Το καταγράφουμε και σας ευχαριστούμε. Σημείο 4. Σας είπα για την αλλαγή των σημείων της σας διάταξης ε, μετά από αίτημα της κυρίας Σάρβου τη συντάκτηρα γνωμοδότη. Δηλαδή το 7 θα το συζητήσουμε μετά το 9. Και έχουμε ε, διερμηνία από και προ ε, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, δανέζικα, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, σουηδικά, ουγγρικά, ε, λιθουανικά, πολωνικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Και σημείο 5. Ανάλυση με θέμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θέση τους στις παγκόσμιες αγορές τροφίμων γεωρικής προέλευσης τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές. Ανταγωνιστική θέση. Έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας κάνει μια παρουσίαση η οποία θα επικεντρωθεί σε ένα πολύ σημαντικό θέμα την κατάσταση των πραγμάτων μετά το ρωσικό εμπάργο καθώς και τις τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις. Θα λάβουμε υπόψη δηλαδή τις εξωτερικές ε, συνθήκες και πώς ε, επηρεάζουν τον αγροδιατροφικό κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον καλεσμένο εμπειρογνώμονά μας, τον κύριο Χωσέ Μαρία Γκαρσία Άλβαρες Κόκκε, από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια της Ισπανίας, που θα μας παρουσιάσει την ε, ανταγωνιστική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στις διεθνείς αγροδιατροφικές αγορές θα μας αναλύσει τους ε, βασικούς παράγοντες της εμπορικής ανταγωνιστικότητας και θα μας υποβάλει και κάποιες ε, συστάσεις στρατηγικής σημασίας. Ως ήθιστε, θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον εμπειρογνώμονά μας για μια αρχική παρουσίαση και θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, κύριε Γκαρσία Άλβαρες, έχετε το λόγο για την παρουσίαση. Έχουμε δυστυχώς λίγο χρόνο, γι' αυτό παρακαλώ να είστε σύντομος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που έρχομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεση αυτή καταρτίστηκε πριν την εφαρμογή του ρωσικού εμπάργου, οπότε το θέμα αυτό δεν καλύπτεται. Δηλαδή, ο αντίκτυπος του ρωσικού εμπάργου δεν λαμβάνεται υπόψη στην έκθεση. Βέβαια, οι εξαγωγές μας προς τη Ρωσία είναι το 10% των συνολικών εξαγωγών. Σας είπα ότι θα ασχοληθούμε περισσότερο με μεσοπρόθεσμα ζητήματα και θα δούμε κάποια, το ιστορικό, θα δούμε την εμπορική συμπεριφορά του αγροδιατροφικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θέση του στην παγκόσμια αγορά. Θα κάνουμε μια μελέτη των προοπτικών, θα ασχοληθούμε με κάποια στοιχεία της ανταγωνιστικότητας, θα αναλύσουμε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις σε συγκεκριμένες αλυσίδες και θα καταλήξω σε συμπεράσματα και σε κάποιες συστάσεις. Ιστορικό. Ξεκινούμε καταρχήν από τη βάση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αγροδιατροφική αγορά. 87% είναι η εξαγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παγκοσμίω και έχει ε, σαφή προσανατολισμό προς συγκεκριμένα ποιοτικά προϊόντα με προστιθέμενη αξία. Βέβαια, έχει και κάποια τροτά σημεία η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλονται κυρίως στον κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς και στην εξατομίκευση μερικών παραγωγικών δομών. Επίσης, στην ανάγκη εισαγωγής μεγαλύτερης καινοτομίας στις αγροδιατροφικές αλυσίδες. Έχουμε ένα επιτελείο εμπειρογνωμόνων από έξι χώρες. Από κοινού κατέρτισαν αυτή τη μελέτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών μελών εξετάσαμε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανταγωνιστικότητας στις παγκόσμιες αγορές και εξετάσαμε το πεδίο εφαρμογή και την επιρροή των πολιτικών, όχι μόνο των γεωργικών πολιτικών, αλλά και των άλλων πολιτικών που επηρεάζουν τον αγροδιατροφικό κλάδο. Τι εννοούμε όταν λέμε ανταγωνιστικότητα. Χρησιμοποίησαμε διορισμούς σαν αυτούς που χρησιμοποιεί ο Πόρτερ υιοθετήσαμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας και μιλήσαμε για έθνη ή ανταγωνιστικούς κλάδους, για κλάδους που προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και ταυτόχρονα επιτρέπουν τη δημιουργία κέρδους, εισοδημάτων για τις σχετικές θέσεις απασχόλησης. Μιλούμε δηλαδή για δημιουργία εσόδων και μάλιστα με βιώσιμο τρόπο. Όταν μιλούμε για ανταγωνιστικότητα, θα μπορούσαμε να θετήσουμε δύο πτυχές. Μία πιο παραδοσιακή πτυχή, ένα πιο παραδοσιακό πρίσμα για το μερίδιο στις, ε, στις παγκόσμιες εξαγωγές. Είναι ένα παιχνίδι μηδενικού ε, αθρίσματος. Ό,τι χάνω εγώ, κερδίζεις εσύ και το αντίστροφο. Μπορούμε όμως ε, να θεωρήσουμε με διαφορετικό τρόπο την, ε, την ανταγωνιστικότητα, με βάση με, υπό τη σκοπιά της παραγωγικότητας ε, που δημιουργεί και εισοδήματα. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να μιλήσουμε για μακροπρόθεσμα στρατηγικές ώστε να έχουμε θετικό άθροισμα, δηλαδή να βγαίνουμε και οι δύο κερδισμένοι, να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία και άρα να έχουμε και οι δύο εισοδήματα από αυτή την δραστηριότητα. Έχουμε σημαντικά θέματα όπως η ποιότητα, η καινοτομία, προέλευση των προϊόντων, η εγκύτητα των αγορών, ακόμη και η παράδοση. Και όλοι αυτοί οι παράγοντε επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. Ποιε μεθόδους τώρα χρησιμοποίησαμε στην έκθεση αυτή, στην ε, μελέτη αυτή. Έχουμε συμπληρωματικέ μεθόδους που δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά συμπληρώνει μία την άλλη. Καταρχήν έχουμε του βασικού δείκτες εμπορικών επιδόσεων ή εμπορική συμπεριφορά. αλλά και ε, συμπεριφορά εξαγωγών αλλά και εισαγωγών, αλλά κυρίω επικεντρωθήκαμε στι εξαγωγέ. Δεύτερη μέθοδο στηρίχθηκε σε μια επιγραμμική έρευνα προοπτικών σε έναν ευρύ κύκλο ενδιαφερομένων από όλη την ε, αλυσίδα διατροφής, 158 ε, εμπειρογνώμονες από 19 χώρες με σημαντική παρουσία και πανεπιστημιακών αλλά και οργανώσεων αγροτών, δημοσίων λειτουργών είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταποιητών, διακλαδικών οργανώσεων, λιανεμπόρων, αλλά και χονδρεμπόρων. Όλοι αυτοί έλαβαν μέρος στην μελέτη. Και τρίτη μέθοδος είναι συγκεκριμένες ε, ε, περιπτώσεις της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων. Αλλά όχι μόνο παραγωγής, αλλά όλων των κρίκων της αλυσίδας που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Ποια είναι τα αποτελέσματα τώρα αυτής της μελέτης. Θα προσπαθήσω να τα απλουστεύσω γιατί έχουμε εθνικά αποτελέσματα, τομεακά αποτελέσματα και εγώ θα περιοριστώ σε συγκεκριμένους δείκτες. Καταρχήν, το μερίδιο σε αγορές εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχαμε μία μείωση τη τελευταία δεκαετία. Περάσαμε το 25% της παγκόσμιας αγοράς μέχρι που πιάσαμε πάτο το 2011 με ένα 15% αλλά ε, είχαμε έκτοτε μία μικρή βελτίωση. Χάσαμε λοιπόν τη βαρύτητά μας στην παγκόσμια αγορά εξαγωγών. Και σε ό,τι αφορά τους, ε, καθαρούς, τους ε, καθαρών εξαγωγών, εκεί έχουμε το εξαγωγικό ε, υπόλοιπο που είχαμε μέχρι το 2012 μία μείωση και μετά μία αύξηση. Πώς όμως ε, θα προσπαθήσουμε να συμβιβάσουμε τα, τα δύο αυτά στοιχεία της εξίσωσης. Είχαμε καταρχήν μία ύφεση στην εσωτερική αγορά, είχαμε μία μείωση της εγχώριας ε, ζήτησης, γι' αυτό και στραφήκαμε προς εξαγωγές. Αυτό δεν είναι καλό μαντάτο. Βέβαια, η κατάσταση διαφέρει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές χώρες είχαν σχετική επιτυχία, όπως ε, οι χώρες Βαλτικής, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία. Άλλες χώρες είχαν ε, σημαντική μείωση της συμμετοχής στις εξαγωγές. Η Δανία, η Ουγγαρία και η Σλοβενία, για παράδειγμα. Και οι υπόλοιπε χώρε βρίσκεται κάπου στη μέση. Πάντω η πλειοψηφία των χωρών μελών είδαν να μειώνεται το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά εξαγορών. Επίσης, ε, διαφορετική η κατάσταση ανάμεσα στους διάφορους τομείς. Καλύτερα τα πήγαν ε, τα κρέατα, το χοιρινό, επίσης απορροκυπευτικά, σιτηρά και λιγότερο ρόδινη ήταν η κατάσταση στην αλευροποιία, στους ελέγχους πόρους, τη ζάχαρη, τα λίπη και τα έλαια. Είχαμε πρόσφατα μία μείωση της ανταγωνιστικότητας ε, στο γάλα γαλακτοκομικά προϊόντα και αντίθετα ηγετική θέση και σχετική άνθηση στα ποτά και κυρίως στον ίνο τα τελευταία χρόνια. Τι μας λένε τώρα οι εμπειρογνώμονες. Μερικοί είναι αισιόδοξοι και άλλοι απεσιόδοξοι. Ποια είναι η αισιόδοξη προοπτική. Η αισιοδοξία υπάρχει ως προς την ποιότητα και το δυναμικό ανάπτυξης ε, του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως κάποια απεσιοδοξία ως προς την ικανότητα που έχει ο αγροδιατροφικός τομέας να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, ιδιαίτερα εν ώψη του 2020, γιατί οι προοπτικές μας φτάνουν μέχρι το 2020. Σε ό,τι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο και πάλι η απεσιοδοξία επικρατεί, για ορισμένους τομείς τουλάχιστον, και οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η εξωτερική ζήτηση είναι ένα τμήμα της λύσης, αλλά δεν είναι αποκλειστική λύση. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την εγχώρια ζήτηση. Επίσης, οι εμπειρογνώμονες ε, περιμένουν βελτίωση της εμπορικής συμπεριφοράς σε όλους τομείς ε, που επλήγησαν ε, πιο σοβαρά από την κρίση. Για παράδειγμα, για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι σχετικά αισιόδοξοι για το μέλλον οι εμπειρογνώμονες. Επίσης, είναι αισιόδοξοι για τα απορροκυπευτικά στη Μεσόγειο, για το ελαιόλαδο, τον Ίνο επίσης από τις μεσογειακές χώρες και στις ε, εξαγωγές σιτηρών είναι αισιόδοξη. Εκεί υπάρχει μια τάση ε, αυξανόμενη διεθνούς ζήτησης εξαιτία τη ανέβρεση επιστημιστική ασφάλεια, οπότε αυτήν την άποψη οι προοπτικέ είναι θετικέ. Τώρα, ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντε ανταγωνιστικότητα πολλοί παράγοντε αναλύονται από την έκθεση. Εγώ θα επιμείνω σε τρία στοιχεία. Το ένα αφορά την ε, γεωργική παραγωγικότητα που είναι ένα τμήμα της αλυσίδα, δεν είναι το σύνολο της αλυσίδα, γιατί υπάρχει το παραγωγικό τμήμα, το, το τμήμα του γεωργού, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία στην αλυσίδα διατροφής. Καταρχήν, η γεωργική παραγωγικότητα έχει περιοριστεί από το κατακαιρματισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Πάνω από 2 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσει είναι κάτω των 2 εκταρίων. Επίσης, περιορισμένε είναι οι προοπτικέ αύξηση εισοδήματο ε, για τις περισσότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη πτυχή. Έχουμε ένα ποιοτικό άλμα προς την, αξι... προς την αλυσίδα αξιών και βλέπουμε μια... Ε, ένα καλύτερο συντονισμό. Μια καλύτερη οργάνωση και συνεταιρισμοί θα ήταν η λύση για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξιών. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τις ε, οργανώσεις των παραγωγών, θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαχειριστική τους ικανότητα. Υπάρχει ένα πρόβλημα διακυβέρνησης στην αλυσίδα, ε, στους γεωργικούς συνεταιρισμούς και στις οργανώσεις παραγωγών. Και επίσης, υπάρχει μια συγκρούση μεταξύ των κανόνων ανταγωνισμού και της διαπραγματευτικής ισχύω των παραγωγών στην αλυσίδα. Ένα τρίτο στοιχείο της ανταγωνιστικότητας είναι η καινοτομία. Εκεί οι πρόσφατες αλλαγές στη γεωρική πολιτική και η αλλαγή του, της εστίασης στην κοινή γεωρική πολιτική δημιουργεί αισιοδοξία για το δυναμικό της καινοτομία ή την ενεργοποίηση αυτού του δυναμικού καινοτομία στο αγροδιατροφικού τομέα. Λέω υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία γιατί δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα. Θα πρέπει φυσικά να ενισχύσουμε την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας μεταξύ των διαφόρων κρίκων της αλυσίδας και μεταξύ των κρίκων της αλυσίδας και του πανεπιστημιακού κύκλου, του ακαδημαϊκού κύκλου, γιατί δυστυχώς ε, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και των πανεπιστημίων. Υπάρχει μια κατακαιρματισμένη γνώση, κάτι που δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις ε, και υποσκάπτει τη θέση της γεωργίας και την ανταγωνιστικότητά τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μια μικρή παρένθεση, δεν θα μακρηγορήσω ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε. Βλέπετε τους πίνακε με τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ε, ένα πίνακα για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 χωρών και εκεί έχουμε το χάσμα πρωτο... παραγωγικότητας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης με 15 χώρες. Η γεωργική παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 60% της αμερικανικής παραγωγικότητας. Αλλά προσοχή, να μην δούμε μόνο το λόγο, αλλά και την εξέλιξη. Η εξέλιξη της παραγωγικότητας στη γεωργία δεν είναι χειρότερη από την εξέλιξη παραγωγικότητα σε άλλου τομεί. Μιλώ για την εξέλιξη, έτσι, όχι για το λόγο. Και από την άλλη πλευρά είχαμε κάποια μικρή γεφύρωση αυτού του χάσματο τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε η συγκριτική εξέλιξη δεν είναι αρνητική. Ούτε είναι και πολύ αρνητικό ο πίνακα ό,τι αφορά τις αποδόσεις των καλλιεργιών. Σε ορισμένα προϊόντα οι αποδόσει στη στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεγαλύτερες, το Ναραβόστο και το Ρίζι για παράδειγμα, αλλά για τα υπόλοιπα δημητριακά, για τα υπόλοιπα εισιτήρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάπως μεγαλύτερες αποδόσεις από, την Ευρωπαϊ... από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε υπάρχει μικρή πιθανότητα για αύξηση του εισόδηματο. Τα τελευταία χρόνια η τελική παραγωγικότητα των παραγόντων έχει αυξηθεί πιο γρήγορα μεταξύ 2001 και 2011 στο Βόρειο Ανατολική Ευρώπη ή στο Νότο από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείε και στον Καναδά από, ή από ό,τι στην Ανατολική Ευρώπη. Βέβαια εδώ έχουμε χώρες ε, και κοινοτικέ και εξοκοινοτικές. Γι' αυτό η συνολική αύξηση ήταν περιορισμένη. Αυτό που μας διαφοροποιεί όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι δημόσιες δαπάνες στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Βλέπουμε σε ένα πίνακα ότι οι δημόσιες δαπάνες και οι αναπτυξιακές επενδύσεις ε, είναι συγκρίσιμες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκεί που μας ξεπερνάνε κατά πολύ οι Ηνωμένε Πολιτείε και ίσως οφείλεται και στους μεγάλους ομίλους που έχουν και στις πολυεθνικές, οι διαφορές ε, είναι στις ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί είναι πολύ μεγαλύτερες στις Ηνωμένε Πολιτείες. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να, κοινοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε περισσότερα δημόσιε δαπάνε, δημόσιε επενδύσει, αλλά να προσελκύσουμε ιδιωτικέ επενδύσει, εκείνε που υστερούμε σε σχέση με τι ΗΠΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, είχαμε μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά στάθη των τιμών. Στα γαλακτοκομικά είχαμε αύξηση επίση τη ζήτηση εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε και το θέμα τη ισχύω στην αγορά των παραγωγών και των βιομηχανιών. Σε ό,τι αφορά το βόλιο κρέα, είχαμε χαμηλή παραγωγικότητα και κερδοφορία και είχαμε και την πρόκληση του Μαρκοσούρ στα, στα απορροκυπευτικά, είχαμε το θέμα της ε, της αγοράς, τα επιχειρησιακά προγράμματα και την ανάγκη πολιτικών πρόληψη των κρίσεων. Στο ελαιόλαδο είχαμε εντυπωσιακή αύξηση σε μη παραδοσιακές ε, χώρες παραγωγής και ανάγκη εναρμόνιση των προτύπων. Ενώ στον Ίνο είχαμε τον ανταγωνισμό μεταξύ του παλιού και του νέου κόσμου και το βάρο το άχθο του κανονιστικού πλαισίου, ιδιαίτερα στον αμπελονικό τομέα. Ποιο είναι ο ρόλο των πολιτικών. Καταρχήν, στον πρώτο πυλώνα. Εδώ έχουμε μία ολόκληρη μελέτη διεξοδική. Διαβάστε την παρακαλώ. Γιατί η επιρροή των πολιτικών, των άμεσων ενισχύσεων και των πράσινων ενισχύσεων μας δημιουργεί ένα σαφές πλαίσιο. Απ' τη μία θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άμεσες ενισχύσεις, οι άμεσες πληρωμές φαίνεται να καθυστερούν σε κάποιο βαθμό τις προσαρμογές ή τα ενάυσματα για μεσοπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, αλλά από την άλλη πλευρά ένα τμήμα, το πιο ευάλωτο τμήμα των Ευρωπαίων παραγωγών εξαρτώνται από τις ε, άμεσες ενισχύσεις, ιδιαίτερα από τις συνδεδεμένες. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα, τεράστιο το δυναμικό του δεύτερου πυλώνα για την προώθηση της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Βέβαια, μας ε, θλίβει η συρρήκνωση του προϋπολογισμού, οι περικοπές ε, του δημοσιονομικού πλαισίου με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις, ε, κάτι που ίσως περιορίσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών. Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές πολιτικές, έχουν σημαντική επιρροή στην συμπεριφορά των διαφόρων τομέων. Οι διμερείς συμφωνίες είναι μια εύχρηστη στρατηγική και ένας εύχρηστος οδικός χάρτης και υπάρχει και ο κίνδυνος ε, ε, με το TTIP, τη Διατλαντική Εμπορική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων. Ίσως ε, μετα, μετακινηθούν ε, οι προδιαγραφές μας προς έναν ελάχιστο κοινό παρανομαστή, δηλαδή ταχθούν υπέρ μιας μεγαλύτερης ελαστικότητας και μιας χαλάρωσης των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τώρα, βιωσιμότητα και κλιματικές αλλαγές. Με βάση τη μελέτη αυτή, ο παραγωγικός τομέας ε, είναι κάπως επιφυλακτικός. Απ' την άλλη, δημιουργούνται ευκαιρίες ε, και δυνατότητα για ανάπτυξη της καινοτομία, που είναι πολύ πιο σημαντικά από τις απειλές. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψετε να μακρηγορήσω. Θα περάσω τώρα στα συμπεράσματα και στις συστάσεις. Τελευταία διαφάνεια. Μία σύντομη ανακεφαλαίωση της μελέτης μας και της ανάλυσης των δικτών καθώς και της μελέτης των προοπτικών που πραγματοποιήσαμε, καθώς και της ανάλυσης των αλυσίδων αξιών. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σχετικά καλή συμπεριφορά του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού κλάδου, αλλά δεν είναι ισορροπημένο σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο ένα τραβάει από τη μια και ο άλλο προ την άλλη. Άλλοι βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά του, ε, άλλοι τη μειώνουν. Υπάρχει πάντω κατακαιρματισμό τη ευρωπαϊκή αγορά, μια φοβερή αποσπασματοποίηση και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα αυτός ο κατακαιρματισμός στην εύρυθμη λειτουργία της αλυσίδας των αξιών. Επίσης, θέλουμε πιο αποτελεσματικούς και λιγότερο γραφειοκρατικούς κανόνες, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαπιστώσαμε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν έρχεται σε αντιπαράθεση ε, με την ε, κοινωνική και εδαφική συνοχή και τη βιωσιμότητα. Το αντίθετο, ενισχύεται από αυτήν. Επίση, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην εγχώρια αγορά. Καλέ οι εξαγωγέ, αλλά και η εγχώρια ζήτηση, οι τοπικέ αγορέ και η εσωτερική ζήτηση είναι σημαντικά θέματα. Εμπορική πολιτική. Καλό τρόπο. Ε, και η στρατηγική προάσπιση τη Ευρωπαϊκή Εμπορική Πολιτική στα διεθνή φόρα είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουμε συνθήκε ίσου ανταγωνισμού παγκοσμίω. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, προάσπιση των ονομασιών προέλευση ε, στα TRIPS, στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ο δεύτερος πυλώνας, να μην γίνει χαμένη ευκαιρία. Βέβαια, από το τύπο ολότελα καλός και δεύτερος πυλώνας, αλλά χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Και επίσης ε, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε εταιρικέ σχέσεις για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Εκεί θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, θα ενεργοποιηθούν οι τοπικές οικονομίες και θα ενισχυθεί και το δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για την συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή της Άγκρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα υποβληθούν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου επιτρέπετε να σχολιάσω αυτήν την μελέτη. Σαφώς και συνεισφέρει η έρευνα αυτή όσον αφορά την γνώση μας για την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Είναι πάρα πολύ λογικά και ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά, ιδιαίτερα αν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση από καθαρός εισαγωγέας ε, προϊόντων στον τομέα της αγροδιατροφικής βιομηχανίας γίνεται ή μπορεί να γίνει καθαρός εξαγωγέας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δούμε πώς αυτά τα στοιχεία και αυτή η ανάλυση θα μας επιτρέψουν να αποκτήσουμε μια ευρύτερη γνώση όσον αφορά την ανάλυση και τα συμπεράσματα για τον τομέα αυτόν. Πρώτον, ο διτός χαρακτήρας μεταξύ μιας ανταγωνιστικότητας που βασίζεται καθαρά στο κόστος, μια ποσοτική δηλαδή ε, ανταγωνιστικότητα σε σχέση με μια ανταγωνιστικότητα που βασίζεται σε ποιότητα. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τα δύο τμήματα αυτά της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να αναλυθούν με μεγάλη λεπτομέρεια έτσι ώστε όχι μόνο να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας αλλά να υπάρξει περισσότερη προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τα οποία παράγουμε, αλλά και στις επιχειρήσεις οι οποίες ενεργοποιούνται στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Δεύτερον, κάτι που αφορά κατά την άποψή μας πάλι την ανταγωνιστικότητα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στο γεγονός ότι μεταξύ 2001 και 2010 μειώθηκε το ποσοστό των εξαγωγών στον τομέα αυτό. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην περίοδο αυτή υπήρξαν αγροτικοί τομείς ε, σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματικά άνθησαν και αναπτύχθηκαν. Αυτό βεβαίως έδειξε ότι η παραγωγικότητα εδώ παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, ανταγωνιστικότητα. Αν κάποιος εξηγήσει ε, αυτά τα στοιχεία διαπιστώνει ότι η μείωση των εξαγωγών έχει σχέση άμεση με την ε, σχέση μεταξύ επιδοτήσεων και εξαγωγών. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις και η ποσότητα αλλά και η αξία αυτών των εξαγωγών ε, αυξάνεται. Πολλές μελέτες, ε, δημόσιες μελέτες δείχνουν ότι αυτό ισχύει σε πολλές περιπτώσεις και στα συμπεράσματα αυτής της μελέτης βλέπουμε ότι οι πληρωμές όσον αφορά τον πυλώνα 1 βελτιώνουν αυτές τις διακυμάνσεις ε, στην ανταγωνιστικότητα και αυτό που πιστεύουμε είναι ότι υπάρχει συμπληρωματικός χαρακτήρας μεταξύ των πληρωμών αυτών μεταξύ του πυλώνα 1 και του πυλώνα 2 των άμεσων πληρωμών και πολύ σωστά οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αυτών των άμεσων πληρωμών και της ε, διακύμανσης της ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει επίσης να δούμε και το θέμα των τιμών, κάτι το οποίο αγνοεί η μελέτη. Δεν θεωρούμε σε καμία περίπτωση ότι οι εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης θα αλλάξουν εάν ληφθεί υπόψη και αυτός ο παράγοντας. Θεωρούμε όμως ότι σε μελλοντικέ μελέτες θα πρέπει σαφώς και ο παράγοντας των τιμών να λαμβάνεται υπόψη. Ευχαριστώ. Εννέα μέλη της Επιτροπής το λόγο. Θέλει άλλος κανείς ε, να συμπεριληφθεί στο κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία είναι δέκατη ενδέκατος κάποιος εθελοντής. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αργότερα και τον Επίτροπο, τον κύριο Τσόλος. Ενάμιση λεπτό στον καθένα γιατί είμαστε πολύ έντεκα. Έχετε 1,5 λεπτό για να υποβάλλετε τις ερωτήσεις και να προλάβει ο καλεσμένος μας να δώσει απαντήσει. Ο κύριος Ντες, 1,5 λεπτό παρακαλώ κύριε Ντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτής της μελέτης. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Πολύ σύντομη ερώτηση ήθελα να σας κάνω. Μιλήσατε για τις περικοπές ε, στον προεπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε για 15%. Μπορείτε να μας πείτε αν το greening ε, αυξάνει το κόστος εδώ και αν μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα από την περιοχή μου, από τη Βαρβαρία όταν βλέπουμε το greening να επεκτείνεται σε κάποιες περιοχές και βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι αφαιρούνται από τους αγρότες 350 ευρώ ανά εκτάριο καθότι δεν πρέπει να επικαλύπτονται οι διάφορες βοήθειες όπως παραδείγματος χάρη αυτές που δίνονται για τα λουλούδια και για την μελισσοκομεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στις ε, παρατηρήσεις της Επιτροπής για, την για τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Έχω την εντύπωση ότι η σημερινή κοινή αγροτική πολιτική μας ε, δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι αγρότες μας με αυτό το θέμα του greening και με τις άμεσες πληρωμές του δεύτερου και του πρώτου πυλώνα και τις περιπτώσεις επικαλύψεων. Ευχαριστώ κύριε Δεκάστρο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Ευχαριστώ για τη μελέτη. Όλα ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα. Έχω μία ερώτηση. Μιλήσατε για παραγωγικότητα. Ε, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι ε, η Ευρώπη γίνεται σημαντικός παραγωγός αγροδιατροφικών προϊόντων με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιο υπολογισμό συγκεκριμένο, αλλά η στρέβλωση του ανταγωνισμού οφείλεται στους διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των γεωργών της Ευρώπης και των υπολείπων. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή της στρέβλωσης. Ε, ανταγωνιζόμαστε σε μια παγκόσμια αγορά, αλλά οι δικοί μας κανόνες είναι πολύ πιο αυστηροί όσον αφορά τα ποιοτικά πρότυπα. Τα θέλουμε αυτά τα ποιοτικά πρότυπα, θέλουμε και την ευζωία βεβαίως των ζώων, οι άλλοι όμω δεν έχουν αυτού του κανόνε. Όλα αυτά επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη. Δεν είναι... Θα ήθελα τη γνώμη σα. Σας ευχαριστώ κύριο Χόισλινγκ. Ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη σας. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ. Πάντα όταν εξάγουμε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Έχω τρεις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, κατά πόσο αυτή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται και βασίζεται στις άμεσες ε, πληρωμές. Ξέρω παραδείγματο χάρη ότι δεν είναι δυνατόν κανένας παραγωγός στον τομέα των γαλακτομικών προϊόντων και του γάλακτος να ε, είναι η παραγωγή του διαθέσιμη και να μπορεί να διατεθεί συγγνώμη, στην ευρωπαϊκή αγορά με αυτές τις τιμές χωρίς δηλαδή τις άμεσες πληρωμές. Κάτι άλλο που ε, θα ήθελα να πω διαρκώς, οι ζωοτροφές γίνονται και λιγότερο ακριβές όταν προέρχονται από τρίτες χώρες. Είναι γνωστό λοιπόν γιατί εισάγουμε αυτά τα προϊόντα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα όταν υπάρχουν αυτά τα πολύ συγκεκριμένα προϊόντα που είναι τόσο πολύ πιο φθηνά και τα εισάγουμε. Τρίτο σημείο, μιλήσατε για τον κατακαιρματισμό της παραγωγής των μικρογεωργών. Ναι, αυτή είναι όμως η κατάσταση. Το θέμα είναι τι προστιθέμενη αξία, τι αξία μένει στην τσέπη του αγρότη, του γεωργού με αυτές τις τόσο χαμηλές τιμές. Κυρία Σανρά. Κυρία Σάνδρα. Sí, gracias. Ευχαριστώ. Ερώτηση στη μελέτη που εκπονήσατε. Υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει υποχώρηση των μικροκαλλιεργητών ε, στο γενικό τοπίο εξαιτία ε, των νέων τάσεων στις εξαγωγές. Ο κύριος Μποβέ. Oui, bonjour. Euh, euh, la question... Καλημέρα σας. Η παραγωγικότητα κατά την άποψή μου δεν είναι σωστή προσέγγιση. Με την έννοια ότι σήμερα οι εξαγωγές σφαιρικά συναποτελούνται από πλεονάσματα. Και αν πάρουμε τα παραγωγή γαλακτομικών, είναι σαφές σήμερα ότι έχουμε μια αύξηση των πλεονασμάτων μεταξύ των τριών μεγάλων ομάδων. Την Ευρώπη, τη ΣΥΠΑ και Νέα Ζηλανδία που θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα κέρδος για τη γεωργία από τις εξαγωγές. Κανένα κέρδος. Και στα συμπεράσματά σας λέτε ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο ισχυροί στη ε, διμερείς μας ε, διαπραγματεύσεις. Μα αυτές οι διμερείς συμφωνίες θα προκαλέσουν ζημιές στην παραγωγή γιατί σήμερα μιλάμε για 10-15% τουλάχιστον του βόηου της Ευρώπης που εμπλέκεται σε αυτές τις συμφωνίες. να βασίσουμε λοιπόν μια στρατηγική πάνω στις εξαγωγές, αυτό δεν φέρνει τη θέμενη αξία για τους παραγωγούς, μόνο για τους αγροδιατραφικούς ε, κλάδους που χρησιμοποιούν τους γεωργούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπέλτερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, ευρωπαϊκής αγοράς. Διαπιστώνω ότι εδώ πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση και συνθήκες ανταγωνισμού. Βλέπω επίσης ότι ο μηδενικός κοινός παρανομαστής έχει επικρατήσει. Αυτό υπονομεύει την οικονομική υγεία των δικών μας παραγωγών. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα κινδυνεύουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες προϊόντων που θα κατακλείσουν την ευρωπαϊκή αγορά χωρίς καμία προδιαγραφή συγκρίση με τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ο κύριος Ευχαριστώ. Απλή ερώτηση. Είπατε στην παρέμβασή σας ότι το, η δύναμη διαπραγμάτευσης των γεωργών περιορισμένη και συχνά παρεμποδίζεται από το δίκαιο του ανταγωνισμού. Θεωρώ συνεπώς ότι η μελέτη σας έγινε κάτω από την προηγούμενη νομοθεσία του 2013. Δεν εντάξατε τίποτα από ό,τι υπάρχει στη νέα οργάνωση της κοινή αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Σλουαζό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για μας τους Γάρους η έλλειψη ανταγωνισμού οφείλεται σε τρεις βασικές αιτίες. Πρώτα απ' όλα τον ανταγωνισμό που υφιστάμεθα από το, λόγω του κόστους μας, που είναι υψηλότερο από τις τιμές ε, πώλησης των ΗΠΑ και της Βραζιλίας. Ε, με το Farm Bill ε, η ΗΠΑ επαν... ξανάβαλε το ελάχιστο επίπεδο και η Ρωσία θα έρθει να ανταγωνιστεί ακόμη παραπάνω στην αγορά. Δεύτερον, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην επόμενη φάση όταν η αγρανάπευση θα αυξηθεί ακόμη παραπάνω. 3-5% και πάμε. Πώς θα συνεχίσει η Γαλλία να εξάγει προϊόντα όπως κρέας, ζάχαρη, πουλερικά, χωρίς επιστροφές εξαγωγικές. Επαναλαμβάνω ότι το κόστος παραγωγής είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Βαζεχόφσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της μελέτης. Αν κατάλαβα καλά, τον τρίτο πίνακα στη σελίδα 34 φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε τα τελευταία 10 χρόνια μεγάλη μείωση από το 23-25% στο 15%. Ε, δηλαδή αποδυναμώνεται η θέση μας ε, στο παγκόσμιο προσκήνιο σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. Και υπάρχει πρόβλημα ε, δικτών ώστε να συγκρίνουμε τη θέση μας στην παγκόσμια αγορά και να κάνουμε ένα επιμερισμό αναχώρα ό,τι αφορά τη γεωρική παραγωγή. Με τα στοιχεία της Ευρωστάτ φαίνεται ότι η Πολωνία είναι σημαντικός εξαγωγές καφέ ή τσαγιού Καμία σχέση βέβαια αυτό με την, ε, με τα, με την πολωνική γεωργία. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ειδικά για τη γεωργική παραγωγή των επιμέρους χώρων γιατί διαφορετικά φτάνουμε σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Γιατί ε, η μελέτη σας λέει ότι είχαμε ε, μεγάλη άνθηση της γεωργίας στις βαλτικές χώρες στην Πολωνία, ενώ λέτε ότι η Ολλανδία έχει πρόβλημα, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα στη Γεωργία μας. Καμία σχέση με τα στατιστικά στοιχεία, γιατί τα στατιστικά στοιχεία πολλές φορές δεν ε, εμένουν στην ε, αμυγός γεωργική παραγωγή μιας χώρας, αλλά ε, επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα. Ναι, όντως. Είναι πολύ πιο εύκολο να ανέβει κανείς από μια χαμηλή θέση από ότι να πέσει από μια υψηλή. Ο κύριος Ρομπέ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν πραγματοποιούνται αυτές τις μελέτες παίρνουμε τα στοιχεία από το παρελθόν βεβαίως. Και όταν έχουμε τη ρωσική κρίση βεβαίως δεν ξέρουμε ακόμη τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Θα θέλαμε να δούμε κάτι για το 2014 και το 2015. Αναφερθήκατε στα μειονεκτήματα στους περιοριστικούς παράγοντες, στις ε, ελλειπείς διαπραγματευτικές ικανότητες των ενώσεων, όμως δεν περιλαμβάνεται συγκρίσεις μεταξύ κρατών στη μελέτη σας. Σε ορισμένες χώρες έχετε πολλές ενώσεις παραγωγών 17-18% των παραγωγών είναι μέλη τέτοιων οργανώσεων. Τώρα στη Λιθουανία είναι μόνο 15%. Αλλού είναι πολύ περισσότεροι. Ε, μήπως πρέπει να ενθαρρύνουμε ένα συνεργατικό σύστημα για την παραγωγή υλικών, βασικών υλικών κτλ. Ε, ίσως αυτό θα ήταν κάτι που θα γινόταν πιο κατανοητό σαν σύσταση. Ίσως Πρέπει επίσης κάτι να κάνουμε στην αλυσίδα των πληρωμών, ε, να διευκολύνουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γουιτάρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Άλβαρες για την παρουσίαση της μελέτης. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα και φυσικά θα πρέπει να εντρυφήσουμε στη μελέτη γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μάλιστα και προλαλήσαντες τις έθεξαν εν μέρη. Είπατε, κύριε Άλβαρες, ότι δεν έχουν μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ η παραγωγή, η γεωργή. Και επίση προβληματίζει το κανονιστικό πλαίσιο του ανταγωνισμού και είναι σημαντικό για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα να είναι καλά οργανωμένη η γεωργή η παραγωγή. Ερωτώ λοιπόν, τι γνώμη έχετε, πώς μπορεί να βελτιωθεί η οργάνωση των παραγωγών και πώς μπορεί να διορθωθεί αυτή η αντιπαράθεση με τους κανόνες του ανταγωνισμού, όχι μόνο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο γιατί υπάρχουν διαφορέ ό,τι αφορά την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών μελών. Και αυτό θίγει την ανταγωνιστικότητα. Επίσης, τι γίνεται με την οργανωτική δομή. Θεωρείται ότι ο συνεταιρισμό είναι μια κατάλληλη μορφή οργάνωση που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των γεωργών. Σα ευχαριστώ. Κύριε Χανιώτη, θέλετε να μιλήσετε πριν τον καλεσμένο μας, τον εμπειρογνωμονό μας. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρία σχόλια σύντομα σε σχέση με τις ερωτήσεις που μας απευθύνεται. Όσον αφορά το greening και το πρόσθετο κόστος του greening σε σχέση με την παραγωγικότητα. Ε, θέλουμε να κρατήσουμε βοσκότοπους εκεί που υπάρχουν. Αυτό δεν επηρεάζει την παραγωγικότητα, τουλάχιστον βελτιώνει την αποδοτικότητα της γης και μειώνει τις εκπομπές. Το greening σημαίνει ποικιλομορφία στα φυτά και επίσης έχει να κάνει και με την EFA. Οπωσδήποτε η EFA είναι πιο περίπλοκη και πιο προβληματική από αυτό που νομίζαμε στην αρχή αλλά η EFA αφορά μόνο ένα με 2% της αεροτριέας γης. Θα συζητηθεί και του χρόνου βέβαια. Χωρίς να αποφεύγουμε να το συζητήσουμε, πρέπει να το βάλουμε στο σωστό πλαίσιο. Οπότε η επίδραση πάνω στην παραγωγικότητα θα είναι περιθωριακή. Άμεσες πληρωμές. το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα δεν έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Έχουμε κάνει επανειλημμένες ε, μελέτες στο σενάριο 2020 είναι μια τέτοια μελέτη. Το διαρθρωτικό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή η γεωργία οικονομικά θα είναι πιο ανταγωνιστική χωρίς άμεσες πληρωμές αλλά θα πληρώσουμε πολύ μεγάλο κοινωνικό κόστος λόγω της εγκατάλειψης της γεωργίας σε ορισμένες ευάλωτες περιοχές, τις πιο ευάλωτες ίσως και γι' αυτό πάντα πρέπει να έχουμε μια ισόρροπη προσέγγιση που να εξετάζει και το περιβαλλοντικό και το οικονομικό και το γεωργικό. Τώρα, το εμπόριο, τι ρόλο παίζει. Αν πάρετε τα δεδομένα θα δείτε ότι ε, η Ευρώπη έχει σταθερό πληθυσμό, αν όχι μειούμενο. Η Ευρώπη έχει μάλλον ένα χαμηλό ή υπερβολικά χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Ε, ο υπόλοιπο κόσμος αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα. Έχουμε φτάσει σχεδόν στην ε, στον κορεσμό στην Ευρώπη. Όσον αφορά το, την παραγωγή τροφίμων, έχουμε υψηλό κόστος παραγωγής λόγω του υψηλού κόστου της γης, διότι είμαστε μέρος του παλιού κόσμου και όχι του νέου κόσμου. Λοιπόν, αν η Ευρώπη δεν χρησιμοποιήσει τις πρόσθετες ευκαιρίες που εμφανίζονται στον υπόλοιπο κόσμο, η Ευρώπη θα χάσει, και με, σε σχέση με τη γεωργία και σε σχέση με την ανάπτυξη και σε σχέση με νέες ευκαιρίε στον τομέα. Πρέπει να προσθέσουμε αξία αυτό που παράγουμε και υπάρχουν συγκεκριμένα συγκεκριμένα παραδείγματα πώς τα έχουμε κατεφάρει τα τελευταία δέκα χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, παρακαλώ έχετε το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πληθώρα ερωτήσεων. Πολύ εύστοχες ήταν ε, και μεστές. Θα προσπαθήσω να τις συμπιλήσω, να τις ομαδοποιήσω και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων αν ε, παραλείψω καμία από αυτές. Με τη μελέτη ακριβώς εντοπίσαμε τους τομείς στους οποίους χρειάζεται μια περαιτέρω ευάθυνση και μια περαιτέρω εξειδίκευση του έργου. Και ε, εκεί φαντάζομαι θα εστιαστούν στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Χανιώτης, συμφωνώ ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε συγκεκριμένα θέματα, πρέπει να εντρυφήσουμε σε ορισμένα από αυτά και στην έρευνα που κάναμε εμείς με τους ενδιαφερόμενους ε, επικεντρωθήκαμε σε δύο πτυχές της ανταγωνιστικότητας και ευχαριστούμε για τη σύσταση γιατί αυτές τις δύο πτυχές ε, μπορούμε να τις αναπτύξουμε περαιτέρω στις μελλοντικέ μας έρευνες και μελέτες. Δεν αποκλείεται άλλωστε ε, οι αλλαγές στις ενισχύσεις τα τελευταία χρόνια να επηρέασαν ε, το μερίδιό μας στις ε, διεθνείς εξαγωγές. Και φυσικά υπάρχει το θέμα της επιπληρωματικότητας των πυλώνων. Ο πρώτος πυλώνας έχει θεμελιώδη ρόλο. Κανένας δεν προτείνει κατάργηση του πρώτου πυλώνα. Το αντίθετο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην αποτελεσματικότητα του δεύτερου πυλώνα. Όταν μιλούμε για περικοπές στο δεύτερο πυλώνα, το πρόβλημα δεν είναι το 13%. Το πρόβλημα είναι ότι το 13% της μείωση, σε συνδυασμό με τα προβλήματα εφαρμογής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για ένα πυλώνα που δέχεται σύγχρηματοδότηση. Και η μισή Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ δινή κατάσταση οικονομική για να μπορεί να συγχρηματοδοτήσει κάποιες δραστηριότητες. Οπότε δεν μιλούμε μόνο για προπολογισμού και για αμυγείς περικοπές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους κανόνες εφαρμογής του πυλώνα αυτού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους μικροκαλλιεργητές, μικροπαραγωγούς, εγώ σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι είναι περίτη άχρηστη η μικροπαραγωγή το αντίθετο. Όταν μιλούμε όμως ότι 6 εκατομμύρια με παραγωγών έχουν λιγότερο από 2 εκτάρια γης, μπορεί να κάνω μια υπεραπλούστευση, γιατί σίγουρα πολλοί από αυτούς ε, ε, επικεντρώνονται σε προϊόντα ποιότητας, σε αγορές που είναι κοντά στον τόπο παραγωγής, μπορεί να συμμετέχουν σε οργανώσεις ή σε συνεταιρισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει τον ε, την ολοκλήρωση αυτή την οργανωτική να την επιδιώξουμε και σε υπερεθνικό επίπεδο. Και όταν μιλούμε για μια παραγωγική βάση όπου αυτοί οι μικροπαραγωγοί έχουν μέσο όρο ηλικία 60 ε, έτη και όταν υπάρχει πρόβλημα κατάρτισης και επιμόρφωσης και μερικές φορές δεν υπάρχει γνώση για το, στις πόλεις για το τι εστί ύπεθρος και τι εστί αγροτική ε, ανάπτυξη, πρέπει να δώσουμε ναύσματα για να προσελκύσουμε μια νέα γενιά γεωργών που θα πάρει τη σκητάλη από τους πιο ηλικιωμένους γεωργούς. Δεν έχουμε ακόμη δώσει αυτά τα ενάυσματα και οι τοπικές αγορές έχουν θεμελιώδη σημασία. Εγώ ουδέποτε δεν είπα ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις εξαγωγές σε Εγώ είπα ότι μειώνουμε τις εξαγωγές μας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή και μάλιστα αυτό ε, είναι συμβατό και με το ε, υπόλοιπο, το καθαρό υπόλοιπο το εξαγωγικό. Και αυτό οφείλεται στην ε, έλλειψη ή στην ύφεση της εγχώριας ζήτησης. Θα πρέπει λοιπόν να μην μας απασχολήσει μόνο η εξωτερική ανταγωνιστικότητα, αλλά η τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Γιατί αυτό δεν υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν και καλύτερη οργάνωση των παραγωγών να έχουμε και τόνωση της εγχώριας ζήτησης και επίσης να δούμε γιατί είναι χαμηλή αυτή η εσωτερική ζήτηση. Και το θέμα, το θέμα της διαπραγματευτικής ισχύως Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμια φόρα. Είδαμε στη μελέτη ότι αυτή η προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών είναι σημαντική. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο, ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που στηρίζεται στην προάσπιση κοινωνικών αξιών, περιβαλλοντικών αξιών Αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να το δώσουμε υπέρ των αξιών μας και στα διεθνή φόρα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για το TTIP για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Και φυσικά λαμβάνοντα υπόψη ότι τα προϊόντα μα πρέπει να είναι υψηλή ποιότητα και προστιθέμενη αξία. Αυτά θα πετύχουμε, αυτέ τι προκλήσει θα τι πετύχουμε με περισσότερη καινοτομία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας όχι μόνο από την κορυφή προς τη βάση, από τους ε, ομίλους και τις πολυεθνικές του μικροπαραγωγούς, αλλά με συνεργασία των διαφόρων ε, φορέων και παραγόντων. Και επίσης ε, να φέρουμε και τους ακαδημαϊκούς κλάδους κοντά στους παραγωγούς, ώστε να εκμεταλλευτούν και την επιστημονική γνώση. Αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί οι εξωτερικές συνθήκες μερικές φορές επηρεάζουν και την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και την λειτουργία της κοινή γεωργικής πολιτικής. Οπότε, όλο και περισσότερο, η γεωργία μας δεν εξαρτάται μόνο από εσωτερικούς παράγοντες, αλλά και από εξωτερικές συνθήκες. Ευχαριστώ λοιπόν το καλεσμένο μας και θα καλωσορίσω τώρα θερμά τον Επίτροπο Τσόλος, που τον παρακαλέσαμε να έρθει σήμερα για μια ανταλλαγή απόψεως ότι αφορά την λειτουργία της ε, γεωργικής πολιτικής, ε, τον απολογισμό του έργου του και τι έγινε τελευταία πενταετία σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Είχαμε πολλαπλές ε, συναντήσεις με τον Επίτροπο, είχαμε μια σειρά ε, συζητήσεων ε, για φλέγοντα και πολλές φορές επίμαχα και επίπονα θέματα. Μιλήσαμε για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής και για μία σειρά θεμάτων. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της κοινή γεωρικής πολιτικής. Έχουμε μέχρι τώρα πάντως συγκεντρώσει αρκετά πλούσια πείρα ως προς το θέμα αυτό και θεωρήσαμε σκόπιμη μια ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Τζόλος, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την ε, παρουσία του εδώ. Μετά την παρουσίαση την αρχική από τον Επίτροπο θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Χρόνο έχουμε μέχρι τις 6.30. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Merci, euh, Monsieur le euh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι η τελευταία μου συνάντηση μαζί σας σαν Επίτροπος Υπεύθυνος για Γεωργικά Θέματα. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα συγκινημένος. Είμαστε εν μέσω των ακροάσεων και θυμάμαι σήμερα πριν από πέντε χρόνια, σχεδόν πέντε χρόνια, όταν ήρθα εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάποιοι μάλιστα από εσάς ήσασταν ήδη εδώ. Μιλήσαμε για τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής, αν θυμάστε. Κάποιοι από εσά ήταν ήδη εδώ και είχαμε πολύ σημαντικές προκλήσεις, οικονομικές, πολιτικές, θεσμικές. Η μεταρρύθμιση της ΠΑΚ σκοπός αυτής της μεταρρύθμισης ήταν να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα, η φορεία της ευρωπαϊκής ε, γεωργίας. Και βεβαίως μιλούσαμε και για τις δημοσιονομικές προοπτικές ταυτόχρονα. Υπήρχε μια σημαντική λοιπόν ε, θεσμική πρόκληση, ήταν η συνθήκη της Λισαβόνας, τη θέση σε ισχύ της, Κάτι που έθετε το Κοινοβούλιο σε μια διαπραγματευτική ισότητα για τα θέματα αυτά. Μάλιστα μου είχατε κάνει την εξής ερώτηση, αν θα υπάρξει επανάσταση ή εξέλιξη στον τομέα της μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η απάντησή μου ήταν μια εξέλιξη της πολιτικής αυτής προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι ότι η μεταρρύθμιση προχώρησε, έδωσε περισσότερα μέσα και εργαλεία στους ε, Ευρωπαίους αγρότες και την ίδια ώρα περισσότερη νομιμότητα θα έλεγα. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το θέμα της διατροφής στην Ευρώπη, το θέμα της αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη για σημαντικά θέματα με επιπτώσεις ε, πολύ σημαντικές για την οικονομία, για τις εμπορικές μας σχέσεις και στον κοινωνικό τομέα. Πριν ξεκινήσει αυτή η μεταρρύθμιση, η κοινή αγροτική πολιτική ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων εντός και εκτός του αγροτικού τομέα το θέμα της διατροφής, το θέμα της υπαίθρου, το θέμα των ε, γεωργών έπρεπε να βγει και εκτός αυτού του γεωργικού τομέα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ευρεία συζήτηση η οποία θα προετοίμαζε το έδαφος αυτής της μεταρρύθμισης. Όπως ξέρετε, το θέμα του greening, καθώς και άλλες αποφάσεις που ελήφθησαν σε πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης, μας βοήθησαν να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Περισσότερη ευελιξία επίσης. 28 κράτη-μέλη με πολύ διαφορετική κατάσταση που επικρατεί για τους γεωργούς μας από τη μία χώρα στην άλλη χρειαζόταν ευελιξία. Αν θέλαμε να παραμείνει η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική πραγματικά κοινή. Κοινή πολιτική λοιπόν με ευελιξία για τα κράτη-μέλη και για τις περιφέρειες των κρατών μελών. Για τις ε, περιφέρειες μας. Όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές, περάσαμε παραδοσιακό όσον αφορά τα κριτήρια όπως ξέρετε οι αποφάσεις είχαν ληφθεί πριν από 20 χρόνια όσον αφορά τον καταμερισμό αυτών των ε, άμεσων πληρωμών. Παραδοσιακές λοιπόν αποφάσεις που είχαν ληφθεί πριν από 20 χρόνια, οι οποίες θα αντικαταστάθηκαν με πιο στοχευμένες αποφάσεις και κριτήρια που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των κρατών μελών. Άμεσες, πληρωμών, άμεσες πληρωμές συγγνώμη, που είναι ένα στοιχείο στήριξης των αποδοχών του εισοδήματος των γεωργών καθώς και την συνεισφορά της εργασίας των γεωργών στις δημόσιες πολιτικές. Αυτό για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον των γεωργών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πολυμορφία της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη τις πιο ευάλωτες περιοχές σε αγορές με πολύ σημαντικές διακυμάνσεις έτσι ώστε να στηρίξουμε τις πιο ευάλωτες περιοχές, τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, τις ορεινές περιοχές να συνεχίσουν να αποτελούν τμήμα της ευρωπαϊκής ε, αγροτικής πολιτικής. Αποκτήσαμε μάλιστα νέα εργαλεία έτσι ώστε να μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σε περίοδους κρίσης για να μπορέσει κάποιος να προσαρμόσει τα προϊόντα του σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς. Βεβαίως δεν μπορούμε εδώ να εγκαταλείψουμε τους γεωργούς μας στο έλεος των αγορών. Αποφασίσαμε λοιπόν να δημιουργηθεί αυτό το απόθεμα κρίσης, καθώς και η ρήτρα έκτακτης ανάγκης, μια γενικευμένη ρήτρα, έτσι ώστε να μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε, να την επικαλεστούμε κάθε φορά που υπάρχει ε, μια σημαντική κρίση, όπως παραδείγματο χάρη αυτή που προέκυψε τώρα μετά από το ρωσικό εμπάργο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σκεφτούμε ότι τέτοιες κρίσεις ή όπως αυτή του 2009 στον γαλακτοκομικό τομέα επιτρέπουν σήμερα στην Επιτροπή να επέμβει, να αντιδράσει με ταχύτητα. Παρόλο που πάντα πρέπει να ακολουθούμε κάποια στάδια στην ε, αντίδρασή μας. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι το κάναμε και για τα όπορο και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα διαθέτουμε νέα εργαλεία, τα γνωρίζετε και νομίζω ότι σαφώς αυτά τα νέα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καλύτερο τρόπο, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους έτσι ώστε για την επόμενη πενταετία να μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε ενώ βλέπουμε ότι οι δημοσιονομικοί πόροι περιορίζονται. Άρα θα πρέπει σαφώς να βελτιώσουμε τον τρόπο που αντιδρούμε και που παρεμβαίνουμε. Όσον αφορά τώρα τον, την ανταγωνιστικότητα, λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού τομέα, παρόλο που όταν μιλάμε για αγροδιατροφικά προϊόντα, Θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο των γεωργών στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Πολλά ακόμα βεβαίως πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρετε, με τη νέα της ανακοίνωση ανοίγει νέες προπτικές για τα επόμενα χρόνια. Έτσι ώστε πραγματικά να ενισχυθεί ακόμα περισσότερα ο ρόλος των γεωργών στην διατροφική αλυσίδα. Το θέμα τώρα της ανάπτυξης ε, της υπαίθρου, σημαντικός παράγοντας ε, για την βελτίωση των συνθήκων στην αγορά εργασίας, οικονομική στήριξη των ε, γεωργών. Η ανάπτυξη της υπαίθρου σίγουρα αποτελεί έναν από τους προσανατολισμούς για τον εξυγχρονισμό της δραστηριότητας ε, στην Ήπεθρο με συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις, στήριξη στις πιο ευάλωτες περιοχές και αυτό που προβλέπεται βεβαίως στον πρώτο πυλώνα με τα μέτρα επέμβασης της αγοράς και τις άμεσες πληρωμές. Συμπληρωματικός χαρακτήρας λοιπόν μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα, έτσι τουλάχιστον τα βλέπω εγώ, συμπληρωματικά εργαλεία και πιστεύω ότι η επόμενη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής σίγουρα θα βοηθήσουν έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη συνοχή μεταξύ αυτών των δύο πυλώνων της κοινή αγροτικής πολιτικής μαζί με άλλα δημοσιονομικά εργαλεία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εδώ αναφερόμαστε σε ανάπτυξη, αναφερόμαστε σε δημιουργίες νέων θέσεων απασχόλησης. Είναι όμως σαφές ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη σύγκληση μεταξύ όλων των δημοσιονομικών μέσων που προβλέπονται στον τομέα αυτών. Εκτός από τις προσπάθειες για την ΚΑΠ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω αυτά τα οποία κάναμε μαζί για να αξιοποιήσουμε καλύτερα την προστιθέμενη αξία και την ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων. Με τον κανονισμό για την ποιότητα που υπογραμμίζει, επικεντρώνεται αν θέλετε στην ποιότητα και ανήκει οι νέες για δίκτυα και για τις ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων όπως τα ορεινά προϊόντα μας δίνει δηλαδή την δυνατότητα να προωθήσουμε αυτά που, αυτό που θα δώσει θέμενη αξία σε ευρωπαϊκά προϊόντα και θα μπορέσει να το προωθήσουμε το προϊόν και στη διεθνή αγορά. Ακόμη θα ήθελα να σας πενθυμίσω τα εργαλεία προώθησης τα οποία εγκαθιδρύσαμε με δυνατότητες ευρύτερης δράσης στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά με κονδύλια τα οποία ήταν πιο ουσιαστικά ώστε αυτά που αποκαλούμε Made in Europe να μπορούν να παρουσιαστούν στις διεθνείς αγοράς, αγορές όπου υπάρχει δυναμικό εξέλιξης με βάση την ποιότητα, την ποικιλομορφία της παραγωγής μας. Ακόμη υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το εξή, η έρευνα και η καινοτομία. Δημιουργήσαμε έναν πραγματικό μηχανισμό στην πολιτική της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και στην ΚΑΠ, ώστε το αποτέλεσμα της έρευνας και της καινοτομίας να φτάνει στη γη, στο επιτόπου και νομίζω ότι αυτός ο μηχανισμός θα είναι βασικός μηχανισμός για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της απόδοσης της ευρωπαϊκής γεωργίας για όλες τις κατηγορίες γεωργών για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και για τις μικρές, για τις παραγωγές που απευθύνονται στην εξαγωγή όπως και για τις παραγωγές για τοπική κατανάλωση. Στο διεθνές επίπεδο θα έλεγα ότι με τα ρύθμιση της ΚΑΠ αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ε, διαπραγματευθήκαμε τις εμπορικές συμφωνίες μας δώσαν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε για να εξασφαλίσουμε την νομιμότητα της ΚΑΠ θυμόσαστε αποφασίσαμε να περιορίσουμε τις εξαγωγικές επιστροφές. Αποφασίσαμε ακόμη στην εταιρική σχέση με την Αφρική να μην χρησιμοποιούμε πλέον τις εξαγωγικές επιστροφές και αυτό το εφαρμόσαμε μονομερός στην Ευρώπη αν και δυστυχώς η οι συνέτεροι μας, οι διεθνείς αν θέλετε, οι άλλες χώρες δηλαδή, δεν, δεν κατήργησαν αυτό το στρεβλωτικό μηχανισμό. Ακόμη, συζητήσαμε και προχωρήσαμε το φάκελο σε σχέση με τις γεωγραφικές επισημάνσεις προχωρήσαμε σε συμφωνία με τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη και έχουμε προχωρημένη συζήτηση με την Κίνα για την αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων των δικών μας στην ε, κινέζικη αγορά. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι τώρα έχουμε συνέπεια μεταξύ αυτού που κάνουμε στην ΚΑΠ και αυτού που πράττουμε στην πολιτική ανάπτυξης και συνεργασίας όταν αναφερόμαστε στη γεωργία και στην διατροφική ασφάλεια. Όσον αφορά τον τρόπο εργασίας, μπορούμε να βγάλουμε κάποια διδάγματα από αυτά τα πέντε τελευταία χρόνια. Η διαδικασία της συναπόφασης κατά την άποψή μου ήταν παραγωγική όχι μόνο για το Κοινοβούλιο για την επεξεργασία της νομοθεσίας αλλά νομίζω ότι με την συμμετοχή του Κοινοβουλίου ε, νομιμοποιηθήκαμε περισσότερο αν θέλετε για την ΚΑΠ και στο επίπεδο της Κομισιόν σαν εκτελεστικός βραχίωνας νομίζω ότι μπορούμε σήμερα να πούμε ότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση και να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας το γεγονός ότι έχουμε ένα πραγματικό πραγματικό δεύτερο εταίρο το Ευρωκοινοβούλιο και πρέπει να προσαρμόσουμε τη μέθοδο εργασίας μας ε, στην ε, πολιτική ιδιομορφία της εργασίας του Ευρωκοινοβουλίου. Και είμαι σίγουρος ότι στην επόμενη ε, επιτροπή αυτό το στοιχείο θα γίνει ακόμη περισσότερο ορατό. Πάλι όσον αφορά τη μέθοδο εργασίας, ε, είχαμε δημόσιες συζητήσεις και συμμετοχή της ευρύτερης κοινωνίας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΚΑΠ και πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος της μεθόδευσης είναι απαραίτητος για την νομιμότητα της ΚΑΠ και όλοι έχουμε να κερδίσουμε βάζοντας στην ευρύτερη δημόσια ατζέντα το θέμα της γεωργίας, της αγροτιάς και των τροφίμων. Μια τελευταία λέξη. Ένα από τα σημαντικά θέματα για το μέλλον, ξέρω ότι είναι για σας, πώς θα εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση που πετύχαμε απλούστερα με λιγότερη γραφειοκρατία. Αλλά και εσείς ζητούσατε περισσότερη ευκαμψία για τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή. Ξέρετε ότι η Κομισιόν κάθε χρόνο πρέπει να αποδώσει λογαριασμό ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με τη διαχείριση των κονδυλίων στην ΚΑΠ. Ε, αν μου επιτρέπετε μία πρόταση λοιπόν θα έλεγα ότι στο μέλλον θα ήταν πολύ χρήσιμο για την ΚΑΠ να έχουμε μία συντονισμένη εργασία μεταξύ της Επιτροπής Γεωργίας και της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, πάντα του Ευρωκοινοβουλίου, ώστε το Ευρωκοινοβούλιο να μιλάει με μία φωνή όταν μιλάμε για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και όταν μιλάμε και για τη σωστή ορθή διαχείριση των κονδυλίων. Γιατί πιστεύω ότι στα μελλοντικά χρόνια ε, θα ληφθούν πολιτικές αποφάσεις όσον αφορά την ορθότητα της διαχείρισης των κονδυλίων και, την, και το ποσοστό λάθους και ταυτόχρονα θα, θα υπάρξει και το θέμα της ευκαμψίας που πρέπει να δοθεί στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες και ε, ακόμη θέλουμε και αποτελεσματικότητα με όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Αυτές τις σκέψεις ήθελα να σας παρουσιάσω ε, δεν αναφέρθηκα περισσότερο για το εμπάργο της Ρωσίας, ε, διότι ξέρω ότι οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες ε, θα σας παρουσιάσουν αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί, αλλά αν υπάρξουν ερωτήσεις, ευχαριστώ να σας απαντήσω. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε πίτροπε. Έχω ήδη 19 ομιλητές. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το κατάλογο. Αλλά ένα λεπτό ο καθένα το πολύ. Άντε, ένα λεπτό και δέκα δευτερόλεπτα. Αλλιώ δεν προλαβαίνουμε. Εξήμιση πρέπει να ολοκληρώσουμε. Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα ο κύριος Επίτροπος και στην κρίση που μας ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε πολλά θέματα συζήτησης αλλά παρακαλώ να περιοριστείτε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτα θα δώσω το λόγο στους συντονιστές. Πρώτα ο κύριος Δες, μετά ο κύριος Δεκάστρο, κατόπιν ο κύριος Χόουσλινγκ, μετά ο κύριος Άγνιου και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο. Θα ήθελα κύριε Επίτροπε να σας πω ότι κανείς δεν αμφισβητεί την καλή σας θέληση, τις προσπάθειές σας να πετύχετε αποτελέσματα. Απ' την άλλη θα έλεγα ότι τα αποτελέσματα στα οποία φτάσατε μετά από αυτές τις προσπάθειες δεν είναι για μένα ικανοποιητικά. Γιατί πραγματικά όσον αφορά την προσπάθεια να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα για θέματα όπως παραδείγματο χάρη της κατεξουσιοδότηση πράξης. Μετά από δύο χρόνια βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη αγροτική μεταρρύθμιση. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ξέρετε αυτό που θέλω να σας πω και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Αν πραγματικά οι γεωργοί, οι αγρότες της Ευρώπης παρακολουθήσουν αυτά στα οποία φτάσαμε, αυτά τα αποτελέσματα, πολύ φοβάμαι και ανησυχώ για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Σας εύχομαι πάντως κύριε Επίτροπε κάθε καλό και σας ευχαριστώ για, τη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, δεν είναι ώρα να κάνουμε απολογισμό όλο πλήρη της ε, προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας. Είχαμε πολλά θέματα, πακέτο γαλακτοκομικού τομέα, ε, δημοσιονομικές προοπτικές, ε, δυσκολίες να βρεθεί μια νέα νομοποίηση για την κοινή γεωρική πολιτική, πιέσεις από όλες τις πλευρές, όλοι ήθελαν κονδύλια για τη γεωργία πλούσιο νομοθετικό πρόγραμμα. Επίσης, ε, μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική και την οικολογική διάσταση από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης, ε, κοινωνική και οικονομική διάσταση της γεωργίας εξίσου σημαντικές. Και η συναπόφαση που εμπλουτίζει τη διαδικασία και μας επιτρέπει να αναζητήσουμε προβλήματα, ε, λύσει τα προβλήματα με ένα πιο δημοκρατικό τρόπο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία και την τελευταία πενταετία. Η κυρία Σάνορα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Κύριε Επίτροπε, όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας ε, και τη θητεία σας που πλησιάζει στο τέλος της, ο γαλακτοκομικός τομέας βυθιζόταν σε μια βαθύτατη οικονομική κρίση. Τώρα φεύγετε και μετά την, όλη τη συζήτηση που έγινε για το πακέτο για το γαλακτοκομικό τομέα και όλη την σφοδρή συζήτηση που είχαμε την τελευταία πενταετία, ο γαλακτοκομικός τομέας πάλι βρίσκεται στο χείλος μιας σοβαρής κρίσης. Διάβασα πριν από λίγο μια Ολλανδική μελέτη που βεβαιώνει ότι η τιμή του γάλακτος θα συνεχίσει να μειώνεται και δεν πρόκειται ούτε ε, σε ένα χρόνο να συνέλθει και να ακολουθήσει μια αναδική πορεία. Εγώ λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να αισθενιστώ την αισιοδοξία σας στα θέματα αυτά. Γιατί δεν αναγνωρίζετε την αποτυχία των μέτρων και του πακέτου στο γαλακτοκομικό τομέα. Επίσης, μία από τις δεσμεύσεις που αναλάβατε κύριε Επίτροπε πριν από πέντε χρόνια ήταν να βοηθήσετε και να στηρίξετε τους ε, μικρούς καλλιεργητές, τους μικρούς παραγωγούς και τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Γιατί αθετήσατε αυτή σας την υπόσχεση. Ευχαριστώ. 30 σας θερμά παρακαλώ. Ε, κατά μισό λεπτό υπερβήκατε το χρόνο σας. Δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχασα ένα κομμάτι από, τις, ε, από τα σχόλια του Επιτρόπου, αλλά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία του. Επισκέφθηκε την περιφέρειά μου ε, ε, υπήρχαν πολλές ανησυχίες και σε σχέση με το greening και με άλλα θέματα υπήρχαν ε, ε, περίοδοι αναταραχών, υπήρχαν εποχές που διαφωνούσαμε με την Κομισιόν και εγώ περισσότερο ίσως από τους υπόλοιπους, αλλά θα ήθελα επίτροπε να σας ευχηθώ καλή τύχη. Αντιλαμβάνομαι ότι, έχει, ότι έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας θα υπάρξουν και πολλές διαφωνίες, ό,τι και αν συμβεί στο μέλλον. Τουλάχιστον πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα μέλλον για τους γεωργούς, ώστε να εξασφαλίσουν μια δυνατότητα επιβίωσης, ότι όλοι μας συμβάλαμε σε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πίτρεπε, Σα ευχαριστώ πολύ εξ ονόματο της πολιτικής μου ομάδας για την εργασία σας, για τις προσπάθειές σας και για τον νέο τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε πλέον με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά θεωρώ επίτευγμα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα της νομιμοποίησης των νέων άμεσων πληρωμών. Θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Σήμερα δεν μου δίνονται χρήματα μόνο επειδή είμαι γεωργός, αλλά επειδή συμπεριφέρομαι και αποδίδω σε σχέση με κάποιες συγκεκριμένες ε, πολιτικές. Το θέμα του greening. Το θέμα του greening, ναι, πάμε προς την σωστή κατεύθυνση. Το θέμα βέβαια είναι ποια είναι τα μέτρα που έχουμε θεσπίσει. Οι πληρωμές ε, θα πρέπει φυσικά να ανταποκρίνονται στους προσανατολισμούς στην νομιμοποίηση αυτής της νέας πολιτικής της μεταρρύθμισης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω το έργο σας να συνεχιστεί από την νέα Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μίλλερ. Κύριε Επίτροπε, θεωρείτε ότι με την μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής προστατεύσατε καθόλου τους μικροκτηνοτρόφους, τους μικρογεωργούς. Εγώ είμαι από μια περιοχή που έχει πάρα πολύ μικρούς, μικρές εκμεταλλεύσεις και το βάρος της γραφειοκρατίας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να αντέξουν πλέον οι μικρογεωργοί και οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν παραδείγματος χάρη γιατί χρησιμοποιούμε εδώ παραδείγματος χάρη διαφορετικούς όρους από τους ε, παραδοσιακούς, παραδείγματος χάρη για τα προϊόντα που γίνονται με ανάμιξη φρούτων, γιατί χρησιμοποιούμε άλλους όρους, άλλες ονομασίες, έτσι ώστε να περιπλέκουμε ακόμα πιο πολύ τα πράγματα. Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι αυτή η γραφειοκρατία πλήττει τους μικρογεωργούς, τους μικρούς, τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Επίτροπε, νομίζω ότι το επίκεντρο της όλης υπόθεσης είναι η απαγόρευση των σπόρων βάμβακα που έφερε το ακριβώς αντίθετο επίπεδο. Δηλαδή για τους μελισσοκόμους τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ δεν θα μπορούσε να, είχε, να είχαμε πετύχει χειρότερο αποτέλεσμα έχουμε ένα, μια σκιά πάνω όλη σα τη θητεία σα χωρίς να υπάρχουν λύσει σε κάποιου τομείς. Τώρα, ε, επειδή ε, ε, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν το προηγούμενο, αλλά δεν μπορούν να καλλιεργήσουν και κάτι νέο, υπάρχουν νέοι κανόνες όσον αφορά τους χώρους οικολογικής εστίασης το μόνο που θα μπορέσουμε να κάνουμε είναι ε, κουράγιο. Ε, Λεόκραμβη. Voorzitter, dank u wel. Commissaris, ik ken u in Nederland als uh, pas sinds het sanctie... Σας ευχαριστώ, κύριε Oké, familie hm, θα μιλήσετε λίγο αργότερα. Ε, καταρχήν η κυρία που είναι δίπλα σας. Κυρία Ρανς Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πενταετία στενής συνεργασίας και μεγάλη συμβολή. Συγχαρητήρια για το συνεργάσιμο και επικοδομητικό σας πνεύμα που συνέβαλε στο να έχουμε μια καρποφόρο συνεργασία. Ε, λάβατε υπόψη και τις ανησυχίες των μεσογειακών χωρών. Είδαμε διαφορά την τελευταία πενταετία στη Μεσόγειο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια χάρη στο συνεργάσιμο πνεύμα σας και στο διάλογο που είχατε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, σας ευχαριστώ για την άμεση αντίδρασή σας στο πρόβλημα που είχαμε με το ρωσικό εμπάργκο. Τον Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα, αλλά καθυστέρησε μετά ένα μήνα ε, για να προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα και Είχαμε ένα μήνα κενό μέχρι να φτάσει στο 165 εκατομμύρια για τα προεκυπευτικά. Αυτή η καθυστέρηση δυσαρέστησε ιδιαίτερα τους γεωργούς. Μήπως τουλάχιστον θα μπορούσαμε να προβλέψουμε αναδρομικό χαρακτήρα των μέτρων αυτών. Νομίζω ότι ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να ολοκληρώσετε με αυτή τη θετική νότα τη θητεία σας. Η κυρία Σλάιερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε πίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Αναφερθήκατε στα οποροκυπευτικά, αναφερθήκατε στο γάλα και στο πρόβλημα με τις κυρώσεις και με το θέμα των ε, κυρώσεων του εμπάργου από μέρους της Ρωσίας. Η κρίση επίσης Κάτι που σίγουρα θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη αντίδραση. Ας μην ξεχνάμε όμως... Ευχαριστώ. Είχαμε ένα πρόβλημα με τη γαλλική διερμηνία. Ο κύριος Καρινόφσκι. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, και εγώ Γιώργος θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την τελευταία πενταετία συνεργασίας. Είχαμε πολύ δύσκολες συνθήκες, πολλαπλές προκλήσεις. Θυμηθήκαμε την κρίση πριν από πέντε χρόνια, το πρόβλημα με το εντεροβακτηρίδιο, η κόλλη, πρόσφατα το ρωσικό εμπάργκο. Πολλές προσπάθειες έγιναν και είχαμε και τη μεταρρύθμιση. Τι άλλαξε την τελευταία πενταετία ε, με τη μεταρρύθμιση που πρέπει να πάσα στιγμή να εφαρμοστεί. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ειλικρίνειά σας γιατί είχατε απαντήσει τότε για τις άμεσες ενισχύσεις και τη διαφοροποίησή τους. Είπατε ότι είναι, ε, είναι μέρος ε, τρόπος εκτός της συνθήκης για επανισορρόπηση κάποιων οικονομικών θεμάτων. Δυστυχώς ε, αυτό είναι αλήθεια και έχουμε ακόμη τη, τα ιστορικά σημεία αναφοράς. Σε ό,τι αφορά το ρωσικό εμπάργο, γνωρίζετε ότι ήταν πολύ αρνητικά αρχικά τα μέτρα για την Πολωνία. Βέβαια, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιες αιτήσει αρχικά που είχε κάνει η Πολωνία που απορρίθηκαν. Αυτό είναι άδικο. Σας ευχαριστώ. Κρατήστε σημειώσεις, ε, κύριε Επίτροπε, μπορείτε να τις διαβεβάσετε και στον διάδοχό σας. Ο κύριος Κούσμινγκ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για το πολιτικό αυτό εμπάργο στη γεωρική παραγωγή εκ μέρους της Ρωσίας, γιατί ήταν ε, ε, πολιτικό αυτό το εμπάρκο που επέβαλε η Ρωσία στα γεωργικά μας προϊόντα. Η αντίδραση όμως της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν ήταν πολιτική. Παρόλο που ισχύει εδώ και δύο μήνες αυτό το εμπάργο και έχει γονατίσει ε, τους γεωργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση μέχρι στιγμής. Ενώ καθημερινά πολλούν τα προϊόντα τους ε, και αναγκαστικά σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι μέχρι σήμερα και χάνουν χρήματα. Δεν θεωρείτε κύριε Επίτροπε ότι η αντίδραση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για την ενεργοποίηση του αποθεματικού με τον αργό αυτό τρόπο ήταν λάθος και πολύ σπασμωδικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βρει άλλα κονδύλια. Και ο τρόπος που επεξεργάζεστε τα αιτήματα των γεωργών δεν είναι και πολύ διαφημής. Μέχρι στιγμής ούτε ένα ευρώ αποζημίωση δεν έλαβαν η Γεωργία, επαναλαμβάνω, που σημαίνει ότι πολύ καθυστερημένα φτάνουν τα κονδύλια. Δεν ήταν λάθος αυτή η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Κύριος Ντόρφμαν. Σας ευχαριστώ. Σε ένα λεπτό δεν είναι εύκολο να πει κανεί ε, όλα αυτά τα οποία αφορούν ε, την ολόκληρη θητεία σας εδώ. Μιλήσαμε για τους ε, γεωργούς, Πιστεύω ότι πετύχαμε πολλά τα τελευταία χρόνια μαζί, το θέμα του πακέτου για το γάλα. Πολλά πρέπει να πω ότι τα φέραμε σε αίσιο πέρας μαζί. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι να δούμε τον απολογισμό όλων αυτών των προσπαθειών. Μιλήσατε για ευελιξία στα εισαγωγικά σας σχόλια. Ίσως το παρακάναμε με την ευελιξία τουλάχιστον αν κοιτάξω εγώ τι γίνεται με τη δική μου χώρα, έχω την εντύπωση ότι μέχρι το 2020, και πολύ λυπάμαι που το λέμε αυτό, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα έχουμε φτάσει σε περισσότερη σύγκληση. Πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες να μειωθεί το χάσμα της ανάπτυξης και πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική που υιοθετήσαμε μας οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Βοτσεχόφσκι. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι αξίζεται συγχαρητηρίων ε, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε τα τελευταία πενταετία με το Ευρωπαϊκό Κοινο... που είχατε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εργαστήκατε άοκνα και υπό δύσκολες ε, πολιτικές συνθήκες. Μειώθηκε ο προϋπολογισμός. Πάντως ε, είναι επιτυχία ότι καταφέραμε να εγκρίνουμε την μεταρρύθμιση. Βέβαια είχαμε πιέσεις από το εμπορικό λόμπι που είναι πολύ ισχυρό στην Ευρώπη και ήθελα να μειωθεί η γεωργική παραγωγή για να αυξήσουν τις εισαγωγές φθηνότερων γεωργικών προϊόντων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε ο κύριος Κούσμιου, δυστυχώ δεν ήταν δέωσα η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιμετωπίσει το εμπάργο. Φαίνεται ότι δεν περιμένατε και εφηνιδιαστήκατε από την αντίδραση. Κι όμως ε, η προσάρτηση της Κρυμαίας έπρεπε να μας είχα προειδεάσει. Αν ήμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι και αν είχαμε λάβει νωρίτερα τα μηνύματα, ίσως ε, θα αποτρέπουμε την εφαρμογή του ρωσικού εμπάργου. Ίσως θα έπρεπε να είχαμε αντιδράσει κάπως καλύτερα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, είμαι καινούριος ευρωβουλευτής. Γι' αυτό και δεν μπορώ να αξιολογήσω το έργο σας την τελευταία πενταετία. Πάντως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησατε στη Λιθουανία. Συζητήσαμε για πολλά θέματα και φυσικά και για το ρωσικό εμπάργο και για την καταβαράθρωση των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης είχαμε πρόβλημα με, τον Αφρικανικό, με την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, με επιζωτίες στα βοηδή. Αντιμετωπίσαμε διάφορες κρίσεις και δυστυχώς μερικές φορές δεν έχουμε την δέουσα αντίδραση και επίλυση των προβλημάτων ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το σύστημα των διακανονισμών δεν λειτουργεί σωστά. Οπότε τον ελάχιστο χρόνο που έχετε μέχρι την ολοκλήρωση της αιτίας σας, σας θερμά παρακαλώ, κάντε κάτι. Ο κύριος Κόλτη. Thank you, uh, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ευχές εσάς, Επίτροπε. Ένα από τα πράγματα που έθεσε τουλάχιστον με μένα και με σίγουρα άλλα μέλη ενδιαφέρον ήταν η επίπτωση που είχαν οι επιθεωρήσεις αγροκτημάτων οι εκμεταλλεύσεων πάνω στους γεωργούς. Δηλαδή αισθάνθηκαν ιδιαίτερα την πίεση πολλαπλών επιθεωρήσεων σε κάποια φάση και η γενική άποψη είναι ότι έχει επιδεινωθεί ε, το καθεστώς επιθεωρήσεων τα τελευταία χρόνια. Όλοι δέχονται βεβαίως την ανάγκη να υπάρχουν επιθεωρήσεις ε, ώστε το, να είναι υψηλή ποιότητα, το τρόφιμο το οποίο, το προϊόν που παράγεται στα αγροκτήματά μας. Μπορείτε να φανταστείτε κανένα μέτρο ώστε να είναι δίκαιο αυτό το μέτρο επιθεωρήσεων και για τους γεργούς και για τους καταναλωτές. Euh, Σήμερα βρισκόμαστε στην Επιτροπή Γεωργίας. Κύριε Επίτροπε, ουσιαστικά αφαιρέσατε την ουσία από την γεωργία, από τον νομέα μας. Βρισκόμαστε υπό διπλή πίεση. Από τη μία η άθλια συνθήκη TTIP και άλλες πιέσεις του διεθνούς εμπορίου και από την άλλη το θέμα του περιβάλλοντος και η επόμενη πενταετία και οι νέες προκλήσεις της κοινή αγροτικής πολιτικής. Πλέον οι γεωργοί δεν μπορούν να αποφασίσουν για τον εαυτό τους και έχουν πληγεί τριπλά σήμερα και από το εμπάργκο από μέρους της Ρωσίας. Αν κοιτάξει κανείς ε, τον προπολογισμό βλέπει σημαντικές περικοπές από το 2000 μέχρι σήμερα. Πώς, κύριε Επίτροπε, θα τα βγάλουν πέρα οι Ευρωπαίοι και οργοί, ενώ οι ανταγωνιστές μας είναι σφοδροί και ανελέητοι. Ο κύριος Νταντά. Αγαπητέ Επίτροπα, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε ε, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πενταετίας αναφέρθηκε ότι οι νότιες χώρες βρήκανε ε, βίκον ους κοντά σας και βεβαίως θα πρέπει να βελτιωθούν και οι συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών σας και της Επιτροπής Γεωργίας αλλά αυτό θα το κάνει ο διάδοχός σας. Ε, ε, ταξιδέψτε παντού στον κόσμο για να δείτε τις εξαγωγές μας. Υποστηρίξετε τα, ε, και αντιληφθήκατε τα συστήματα της γεωργίας των άλλων μεγάλων χωρών. Τι διδάγματα βγάζετε για την ευρωπαϊκή γεωργία. Ευχαριστώ. Ο κύριος... Η κυρία Δελάης. <laughs> Δεν πειράζει, δεν πειράζει, λέει η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, είμαι νέα βουλευτής, αλλά είμαι και παραγωγός λαχανικών. Πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος που αντιδράσατε με το εμπάργο της Ρωσίας, έστω και αν θεωρηθεί ανεπαρκής από συναδέλφους, οπωσδήποτε ήταν καλύτερη από τις πρώτες κρίσεις που ε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το τομέα. Έχω ένα ερώτημα. Έχουμε ανάγκη σήμερα να βρούμε νέες αγορές για κάποια προϊόντα, κάποιους τομείς προϊόντων. Και χρειαζόμαστε προώθηση. Ε, θεωρώ ότι είναι άδικο και συμφωνώ με τους άλλους παραγωγούς ότι πρέπει να συγχρηματοδοτήσουμε κατά 50% τον προϋπολογισμό για την προώθηση. Λόγω της προέλευσης αυτής της κρίσης πιστεύω ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να βρει άλλους τρόπους χρηματοδότησης αντί να ζητά από τους παραγωγούς να ε, συγχρηματοδοτήσουν την αναζήτηση νέων αγορών. Λόγω του εμπάργου πάντα. Ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των αμελητών μας. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο παρακαλώντας τον να απαντήσει. Α, η κυρία Μαγκίνες ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα κύριε Επίτροπε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά, σας βρήκα συνεργάσιμο πάντα και σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Ιρλανδία στην αρχή των συζητήσεων μα είπατε λόγια σοφά, τα οποία δεν έχουν πει άλλοι και πρέπει να ακούσουμε αυτό που είπατε για συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Οι ανησυχίες για τις επιθεωρήσεις ε, ε, υπάρχουν και αυτές και αντιλαμβάνομαι και το σχόλιο σας για ανάγκη συνεργασίας με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να μας πείτε ποια είναι η κληρονομιά σας σε σχέση με τη Γεωργία και τι πιστεύετε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν πετύχει. Έχουν διατυπώσει πολλέ επικρίσεις και για την εφαρμογή του greening ε, και νομίζω ότι υπάρχουν δύο θέματα που μπορούμε να βελτιώσουμε στην απόφαση. Δέσμευση με την Κομισιόν πριν συντάξετε όμω μια πρώτη πρόταση και μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. Ευχαριστώ κυρία Κέστιγκερ, αλλά η τελευταία παρακαλώ. Πολύ πολύ σύντομα όσον αφορά το θέμα της Ρωσίας ε, συζητήσαμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο για τις κυρώσεις. Μπορώ να σας ε, κάνω όμως μια άμεση ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν κάποια μέσα από τον προπολογισμό για όλους αυτούς τους γεωργούς οι οποίοι δεν φταίνε τίποτα για την κατάσταση που έχει προκληθεί με την Ρωσία και ευελπιστούν να υπάρξει κάποια στήριξη από μέρους του προπολογισμού. Όσον αφορά την επιπλέον γραφειοκρατία, και εγώ πραγματικά θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Εάν συνεχίζατε σήμερα, κύριε Επίτροπε, σε αυτή τη θέση, τι άλλο θα κάνατε ή τι θα κάνατε διαφορετικά. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Όλα είναι ακόμη δυνατά. Είναι πολύ νέος ο Επιτροπός μας. Έχει καιρό. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε σε κάποια άλλη ευκαιρία, ίσως άτυπα, ανεπίσημα, να ξανασυζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Με ρωτήσατε τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι είναι ορθό να αφήσω τον επόμενο επίτροπο να απαντήσει σε αυτό. Εγώ έκανα ό,τι νόμιζα ότι έπρεπε να κάνω, ας αφήσουμε τον διάδοχό μου, ο οποίος θα έρθει με νέες ιδέες, νέες προτάσεις και δεν νομίζω ότι εγώ πρέπει να δώσω αυτή τη στιγμή τη δική μου άποψη. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας, αλλά θεωρώ ότι ο νέος επίτροπος, ε, ο κύριος Χόγκαν, έχει και την εμπειρία, αλλά η χώρα από την οποία προέρχεται σίγουρα θα τον εμπνεύσει και θα έρθει εδώ με νέες προτάσεις και πολύ ε, χρήσιμες ιδέες. Αναφερθήκαμε λοιπόν στα προβλήματα αυτής της μεταρρύθμισης, τις δυσκολίες και τις αδυναμίες της. Τα τρία θεσμικά όργανα έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Εγώ σαφώς και μπορώ να στηρίξω και να υπερασπιστώ την αρχική μας πρόταση, αλλά υπήρξε διόρθωση, προσαρμογή αυτής της ε, πρότασης και το αποτέλεσμα στο Λουξεμβούργο ήταν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης αλλίωσε την αρχική πρόταση της Επιτροπής, έτσι κι αλλιώς έπρεπε να το δεχτούμε και να το στηρίξουμε. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή ε, διαδικασία και αυτό που είναι πολύ σημαντικό πέρα από την προσωπική μου άποψη είναι να δεχτούμε ότι μια δημοκρατική διαδικασία οδηγεί σε ένα συμβιβαστικό αποτέλεσμα να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Σαφώς και πάντα μεταξύ της αρχικής μας πρότασης και της τελικής τα πράγματα πολλές φορές αλλάζουν, περιπλέκονται θελήσαμε να λάβουμε υπόψη μας τις προσδοκίες και τις προτάσεις όλων ή των περισσότερων. Τις ενσωματώσαμε στην διαπραγμάτευση. Θεωρώ προσωπικά και το έχω πει εξάλλου, μετά από την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής, ότι μετά από ένα χρόνο εφαρμογής και υλοποίησης πολλά θα πρέπει να βελτιωθούν. Είναι κάτι το καινούριο, είναι καινούρια πολλά από τα στοιχεία αυτής της μεταρρύθμισης, καινούρια για όλους και θεωρώ ότι εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη βελτίωση. Θεωρώ όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταστραφεί η έννοια του greening, καθότι πρόκειται για μια επιλογή η οποία δεν είναι απλώς ένα πολιτικό τέχνασμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε τι γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε ότι διαρκώς αναφερόμαστε στην ανταγωνιστικότητα και στην αηφορία της γεωργίας. Δηλαδή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερους πόρους. Αυτή είναι η τάση και θεωρώ ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και σε αυτούς όλους τους τομείς έχουμε αναλάβει ηγετική θέση. Πολλά πρέπει να βελτιωθούν, όμως το γεγονός ότι επιλέγουμε μία πιο αποτελεσματική γεωργία η οποία λαμβάνει υπόψη της οικονομικά στοιχεία, κοινωνικά στοιχεία, την σωστή διαχείριση των πόρων είναι κάτι που σαφώς θα ακολουθήσουν όλες οι χώρες από εδώ και το εξή, όχι μόνο η Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε βεβαίως είναι να μειώσουμε στο ελάχιστο το γραφειοκρατικό άχθο για τους γεωργού μας. Και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε τα πλεονεκτήματα αυτής της γεωργίας. Αυτό που είπατε, κύριε Άγνιου, είναι πολύ σωστό. Ότι δηλαδή θα συνεχίσετε την καλλιέργεια κάποιων προϊόντων επειδή θεωρείται ότι αυτά τα προϊόντα είναι κατάλληλα και όχι επειδή κάποιος επίτροπος τσόλος ή άλλος πήρε αυτή την απόφαση. Και έχετε δίκιο. Κυρία Μίλλερ, αναφερθήκατε στους μικρούς γεωργούς, τις μικρές εκμεταλλεύσεις, αν προστατεύονται σήμερα περισσότερα. Δεν ξέρω, δείξτε μου μια άλλη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής που λαμβάνει υπόψη της τόσο πολύ την θέση των ε, μικροκαλλιεργητών, των μικρών εκμεταλλεύσεων σε δύσκολες και ορεινές περιοχές τον τρόπο παραδείγματος χάρη που δίνονται πλέον οι άμεσες ε, επιχορηγήσεις. Νομίζω ότι σήμερα στην κοινή αγροτική πολιτική διαθέτουμε εργαλεία έτσι ώστε να στηρίξουμε τους ε, μικρούς γεωργούς για την παραγωγή κοινών αγαθών, αγαθών για όλη την κοινωνία. Όταν αναφερόμαστε λοιπόν σε αυτή τη νέα μεταρρύθμιση, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυξάνεται το γραφειοκρατικό άχθος για τους ε, μικρούς γεωργούς. Ακριβώς το αντίθετο θα γίνει με το νέο σύστημα για τις άμεσες πληρωμές, και με το θέμα του πώς εφαρμόζεται το σύστημα του greening για τους μικρογεωργούς. Κύριε Ντοντά, με ρωτήσατε κάτι, αλλά διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα τέχνασμα πίσω από την ερώτησή σας. Τι θα γίνει με όλα αυτά τα ταξίδια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πραγματικά θεωρώ μετά από πέντε χρόνια σε αυτή τη θέση ότι η ευρωπαϊκή γεωργία είναι πιο ανταγωνιστική σήμερα. Πολλά πρέπει να κάνουμε όταν μιλάμε για την ποιότητα, όταν μιλάμε για την ποικιλομορφία των προϊόντων μας. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί από άλλες περιοχές του κόσμου. Θέλουμε να ενισχύσουμε τους Ευρωπαίους γεωργούς και καλλιεργητές. Θέλουμε να στηρίξουμε τα προϊόντα μας. Κάποιος είπε ότι οι Ευρωπαίοι γεωργοί δεν μπορούν πλέον να αποφασίσουν για τις τύχες τους και ότι δεν θα είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουν την εντατική καλλιέργεια, την άκρατη παραγωγικότητα άλλων περιοχών του κόσμου. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία εμπεριέχει εκτός άλλων χαρακτηριστικών και μια μεγάλη προστιθέμενη αξία. Είμαστε ο πρώτος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων στον κόσμο. Εξάγουμε προστιθέμενη αξία, όχι όγκο. Όσον αφορά την αξία των προϊόντων μας δηλαδή, είμαστε ο πρώτος εξαγωγέας. Εξάγουμε προϊόντα, εξάγουμε τεχνογνωσία, εξάγουμε ποικιλομορφία και εξάγουμε παράδοση. Και βεβαίως, αν αποφασίσουμε να απομονωθούμε σε έναν κόσμο που βρίσκεται εν εξελίξη, δεν νομίζω ότι θα είναι προς όφελος των Ευρωπαίων γεωργών. Ίσως θα μειωθούν οι εισαγωγές μας με αυτόν τον τρόπο, αλλά σίγουρα θα μειωθούν και οι εξαγωγές με τον ίδιο τρόπο, θα μειωθούν οι θέσεις απασχόλησης στον τομέα της αγροδιατροφικής αλυσίδας, αλλά και στην γεωργία. Αυτή η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων μας ουσιαστικά προέρχεται από την παράδοση, από την επιστήμη, από την καινοτομία των Ευρωπαίων γεωργών. Σίγουρα η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να δώσει σε όλους ευκαιρίες, σε μικρές εκμεταλλεύσεις, σε μεγάλους παραγωγούς, σε ορεινούς παραγωγούς. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προστατεύσουμε στο μέλλον. Αλλά μία κοινή αγροτική πολιτική η οποία θα προβλέπει κοινούς κανόνες για όλους έτσι ώστε να είναι πιο απλή, δεν νομίζω ότι θα μας οδηγήσει στο επιθυμητό αποτελέσματα. Θα χάσουμε την ποικιλομορφία μας και θα χάσουμε και το πνεύμα των ευρωπαϊκών συνθήκων όταν ιδρύθηκε η κοινή αγροτική πολιτική στην αρχή. Σήμερα είμαστε 28. Πρέπει να δείξουμε καινοτομία, δυνατότητα προσαρμογής έτσι ώστε να παραμείνει κοινή η αγροτική μας πολιτική λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές και την ποικιλομορφία στην Ευρώπη. Τελειώνοντας, θα αναφερθώ στην κρίση, στο εμπάργο της Ρωσίας. Η αντίδρασή μας ήταν άμεση μόλις συνειδητοποιήσαμε τι συνέβαινε στη Ρωσία. Κύριε Βορτζενχόφσκι, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε κάτι καλύτερο. Πώς θα ξέραμε ποια προϊόντα θα επιλέξει η Ρωσία με το που συνειδητοποιήσαμε τι απόφαση θα έπαιρνε η Ρωσία και εδώ απαντάω και στην κυρία Γκαρσία με το που συνειδητοποιήσαμε την απόφαση της Ρωσίας αντιδράσαμε άμεσα ακόμα και αν αυτή η αντίδραση για κάποιους έφτασε τέλος Αυγούστου. Η απόφασή μας ήταν 18 Αυγούστου, ενώ η Ρωσία αποφάσισε το εμπάργο 7 Αυγούστου. 10 μέρες αργότερα το μέτρο τέθηκε σε ισχύ. Γιατί δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε όλους τους παραγωγούς από την Πολωνία και από άλλες χώρες. Γιατί χρειάζεται ένας συγκεκριμένος τρόπος να υλοποιηθεί αυτό το μέτρο δεν μπορούμε τόσο σύντομα να εξακριβώσουμε την ορθότητα των στοιχείων που μας στέλνουν όλοι οι παραγωγοί. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική δράση, χρειαζόμαστε την ε, ειλικρινή στάση των κρατών μελών και των αρχών τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε δίκαιοι με τους γεωργούς μας. διότι εμείς καλούμεθα να διαχειριστούμε αυτούς τους πόρους και είμαστε υπόλογοι, όπως ξέρετε, για τα κονδύλια τα οποία θα διαθέσουμε. Είδαμε πολλές φορές, παραδείγματος χάριν, αιτήματα τα οποία δεν ακολουθούσαν τους ε, κανόνες. Αυτό όμως δεν είναι δουλειά τελικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε εάν δεν υπάρχει αίτημα βάση των κανόνων. Η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να εφαρμόσει τα μέτρα που έχουν θεσπίσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Όπως ξέρετε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν το πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτοί οι νέοι κανόνες. Μας δίνεται κάποιος χρόνος επιπλέον. Μέχρι τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον παλιό κανονισμό που προβλέπει την συγχρηματοδότηση κατά 50%. Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Μαγκίνες αναφέρθηκε στις κατεξουσιοδότηση πράξης, λέγοντας ότι ίσως θα πρέπει να διδαχτούμε από την εμπειρία μας στον τομέα αυτό. Εγώ λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώς και θα πρέπει να δει πώς λειτουργήσε αυτή η διαδικασία συναπόφασης. Και το ίδιο θα έλεγα και για τον τομέα των κατεξουσιοδότηση πράξης. Θα πρέπει δηλαδή, πράξεων, συγγνώμη, θα πρέπει δηλαδή η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτήν την εξουσία, αν θέλετε, που της δίδεται για να τηρήσει τα κείμενα και τις προϋποθέσεις. Την ίδια ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι τίποτα πέρα από το βασικό κείμενο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ε, εν τέλει. Σίγουρα όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας, για το ανοιχτό σας πνεύμα. Εγώ προσωπικά έμαθα πολλά συνεργαζόμενος μαζί σας. Σίγουρα θα παραμείνω κοντά στον γεωργικό τομέα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και σίγουρα μέσω αυτού του τομέα ή μέσω της πολιτικής μας δράσης θα μπορέσουμε να έχουμε και άλλες επαφές στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, ήταν δύσκολα και ενδιαφέροντα χρόνια και για σας και για μας αλλά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή Γεωργίας ε, είμαστε συναρμόδιοι και συνυπεύθυνοι ε, για να αντιμετωπίσουμε τέτοια θέματα όπως μας ε, ανέθεσε η συνθήκη της Λισαβόνας. Ήταν πολύ το έργο σας, δύσκολο αλλά ισορροπημένο και μεστό. Μερικά θέματα δεν εξαρτώνται από εμά, εξαρτώνται και από τους εξωτερικούς παράγοντες και συνθήκες. Η κατάσταση αλλάζει. Σίγουρα θα προβούμε σε μια αξιολόγηση όλης αυτής της περίοδου και θα αποκομίσουμε πολλές εμπειρίες και από τις κατεξουδόντες πράξεις. Έχουμε πολλά να διδαχτούμε και διδαχτήκαμε ήδη πολλά από όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτά τα συναρπαστικά χρόνια. Συνεργαστήκαμε με αίσθηση ευθύνη και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και απέναντι στους Ευρωπαίους Γεωργούς και απέναντι στην Ευρώπη ολόκληρη. Σας ευχαριστώ θερμά, σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή τύχη και είμαι βέβαιος ότι θα ξανασυναντηθούμε. Γιατί είναι τεράστια η πείρα που συγκεντρώσετε και πιστεύω ότι μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και στο μέλλον για τη Γεωργία. Σας ευχαριστούμε θερμά, θερμά ευχαριστώ από όλα τα μέλη της Επιτροπής και σας εύχομαι καλή επιτυχία δύο πληροφορίες οργανωτικές. Σε λίγο έχουμε κοινή συνάντηση στην αίθουσα 5G3, στην οποία θα λάβει μέρος και ο Επίτροπος και θα έχουμε εκθέσεις για τα Δυτικά Βαλκάνια και την προετοιμασία τους ε, για την ενταξιακή προοπτική. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας προσκαλούμε στην αίθουσα 5G3 μέσω μετά το πέρα συνεδρίαση στην ε, παρουσίαση για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο κύριος Άντριο θα είναι ο πρόεδρος και συμμετέχει και στο Κογκρέσο των Ευρωπαίων Γεωργών. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και πάλι θερμά τον Επίτροπο. Γεια σας.